Uh, Συνάδελφοι, τσακ, τσακ, τσακ. Μήπως να αρχίσουμε. Με το σημείο 1, δηλαδή έγκριση της ημερησίας διάταξης. Τη αιτήση του κυρίου Ομάρτζη δεν θα συζητήσουμε το θέμα του σήμερα. Γι' αυτό αρχίζουμε αργότερα. Υπάρχει βέβαια αναμετάδοση στο διαδίκτυο και πρέπει να ξέρουν οι βοηθοί και οι κοινοβουλευτικοί ότι μπορεί να χρειαστεί να επιταχύνουμε τη δουλειά μας ειδοποιήστε όσους λείπουν να έρθουν κι αυτοί. Εγκρίνεται φαντάζομαι η μερίσια διάταξη. Τώρα περνάμε στο 2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της, των δύο συνεδριάσεων του Νοεμβρίου. 18 και 28 και ως συνήθως αν δεν ακουστούν ή εκφραστούν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα θεωρηθούν εγκριθέντα τα πρακτικά. Σημείο 3. Οι ανακοινώσει της Προέδρου. Οι αποφάσεις των συντονιστών θα ανακοινωθούν εν καιρό το δέοντι και εν ευθέτω χρόνο. Δεν έχω άλλες ανακοινώσει. Τέσσερα έχει ακυρωθεί. Πέντε Η πρώτη κατεξουσιοδότηση πράξη που θα εξετάσουμε και με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Διοντολογία για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Πρέπει να σας ξαναπώ ότι αυτή η κατεξουσιοδότηση πράξη υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο σε όλες τις γλώσσες στις 7 Ιανουαρίου. Δηλαδή, οι δύο μήνες που διαθέτουμε για να εκφράσουμε αντιρρήσεις λίγουν στις 10 Μαρτίου. Και αν θέλουμε να εκφράσουμε αντιρρήσεις πρέπει να εγκρίνουμε ψήφισμα που να περνάει από την νομισμένη διαδικασία. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να μην εκφράσουμε αντίρρηση. Θα δούμε σήμερα στη συζήτηση αν μπορούμε να εγκρίνουμε και την αίτηση της Κομισιόν να ακολουθήσουμε την διαδικασία μη αντίρρησης. Αρχίζει η συζήτηση με πρώτο πρώτο τον εκπρόσωπο της Κομισιόν που θα μας κάνει μία παρουσιασούλα. Ορίστε Νικόλαε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πω για το ιστορικό πλαίσιο δύο λόγια. Αυτή η εταιρική σχέση είναι μια βασική αρχή της πολιτικής της συνοχής και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ βασικό συστατικό για την συνταγή επιτυχίας της πολιτικής αυτής. ούτως ώστε έτσι κανείς να ιδιοποιείται ούτως υπήρχε προγράμματα και να εξασφαλίζει ότι θα υπάρχουν αυτοί, αυτά τα σημερινά συστατικά, ε, οπότε έχουμε ε, αυτό το σχέδιο την πρόταση κανονισμού για την κωδικά βιοντολογίας και έτσι να έχουμε τις αξιολογήσεις και η εμπειρία μας ε, μας έχει φανερώσει ότι αυτό είναι χρήσιμο, συστατικό χρήσιμη αρχή και βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει, υπάρχουν διάφορες παραλλαγές και για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει να καλύψουμε διάφορα θεσμικά πλαίσια, παραδόσεις, ε, δυνατότητες των εμπλεκομένων. Οπότε και έτσι να υπάρχει πραγματική αυθεντική βούληση για την επιτυχία. Οπότε γι' αυτό και έχουμε τάξει κάποια ελάχιστα πρότυπα να υιοθετηθούν οι άριστες πρακτικές για όλες τις περιφέρειες και για όλα τα προγράμματα. Έχουν πάνω σε όλα αυτά τα δύσκολα ζητήματα κατά τις ε, διαπραγματεύσεις. Κάποιες κοινέ διατάξεις εγκρίθηκαν ούτως ώστε να έχει την αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει την κατεξοδότηση πράξη με το πράσινο δός που έδωσε το Κοινοβούλιο όσον αφορά τι μέτρων. Λέει ο οργανισμό ότι θα πρέπει μέχρι το 8 Τετάρτο αυτό να έχει εγκριθεί και όπω ε, και εμεί στι ε, 7 Πρώτου το είπαμε. Σε εσά, Πρόεδρε, και θεωρούμε ότι είναι υψίστη προτεραιότητα. Και αυτό διότι ήδη Υπάρχει μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη σημασία αυτό στα πλαίσια των εταιρικών συμφωνιών και των σχετικών προγραμμάτων. Πρόκειται για μια διαδικασία συνεχεία, το βρισκόμαστε στα τελευταία στάδια και θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει η κοινοποίηση της χρησιμοποίησης πράξης όσο γίνεται συντομότερα παρακάτω. απλουράς περιεχομένου. Ακολουθήσαμε αυτές όλες τις ε, ενδελεχείς διατάξεις όπως το Κοινοβούλιο στο άρθρο 5 για τον κανονισμό των κοινών διατάξεων και πρώτα πρώτα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι τον εντοπισμό των εταίρων πρώτα πρώτα είναι αυτή η έννοια των οργανισμών ομπρέλα διότι η πιο δόκιμη εταίρη η πιο αντιπροσωπευτική. Ε, λαμβάνονται υπόψη για αυτή την εταιρική συμφωνία για να καλύψουμε τα κρατημέλη και να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την προαναφερθήσα έννοια των οργανισμών ομπρέλα και έτσι να καλύψουμε όσο γίνεται περισσότερους εμπλεκομένους σε ένα και μόνο πλαίσιο. Να επομένως μία έννοια η οποία δεν καλύπτει από κάποιον ορισμό που έχει δοθεί αλλά εξηγείται. Εξηγείται και χρησιμοποιούμε αυτή την έννοια και βέβαια σε κάθε κράτο μέλο αυτό επιδέχεται άλλη ερμηνεία, άρα νομίζω τα πράγματα είναι σαφή. Εδώ επίσης υπάρχει σαφή μνήμα τη Territorial Cooperation. Και εδώ έχουμε το EGTC, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την εταιρική σχέση και αυτό έχει να κάνει και με τις μακροπεριφυρακές στρατηγικές. Καλές πρακτικές, οι βασικές έννοιες καλύπτουν την διαδικασία της διαβούλευσης, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το Κοινοβούλιο έχει τα στοιχεία που χρειάζεται και εγκαίρως. Και ότι σε αυτή την συμφωνία και στο πρόγραμμα το κράτος μέλος καλύτερα να εξηγήσει πώς συμμετέχουν κάθε φορά οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με το άρθρο 5. Έχουμε τους σχετικούς κανόνες για την Επιτροπή, την Επιτροπή, την Εποπτική, η οποία ε, συμμετέχει και εξασφαλίζει την ε, αποτελεσματική λειτουργία. Επομένως, εδώ δεν εξαντλούνται οι κανόνες, απλώς αναφέρουμε ποια είναι τα συστατικά, ούτως ώστε να έχουμε ένα σημείο αναφοράς και να μπορούμε να επικαλεστούμε την καλή πρακτική. Επίσης, εμπλέκονται οι εταίροι στη λειτουργία του προγράμματος, με τις προτάσεις, με την εποπτεία, με την αξιολόγηση και Έχουμε εδώ και την έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων που αναφέρεται. Ε, τώρα, στον με τις δυνατότητες, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι διαχειριστικές αρχές χρησιμοποιούν τους πόρους της τεχνικής αρρωγής όπου χρειάζεται. Και εδώ επιβάλλεται να εξετάσουν αυτές οι αρχές το αν χρειάζονται την τεχνική αρρωγή. Και αν τη χρειάζονται, την επικαλούνται και συνεχίζουν. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Εντροπή έχει το ρόλο του να διαδώσει τις σωστές πρακτικές και έχει δείξει η εμπειρία ότι έτσι υπάρχει ο κοινός τόπος της ανταλλαγής των ε, σωστών πρακτικών και αυτό γίνεται σε θελοντική βάση πλευρά τη Επιτροπή. Εξαρτάται κάθε φορά ποιοι είναι οι εταίροι. Έχουν τον κώδικα διοντολογία, οι επιβάσει των διαβουλεύσεων και αυτέ οι διαβουλεύσει ε, έχουν κρατήσει πολλού μήνε. Και αυτά τα λέει το άρθρο 5. Ε, ε, αναφέρονται λεπτομέρειε, οι σκοποί, οι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν και έτσι οι εταίροι έχουν σε όλε τι περιφέρειε, σε όλα τα κράτη-μέλη στη διάθεσή τους αυτά τα οποία χρειάζονται για τα προγράμματα. Τώρα, ένα άλλο θέμα, το είναι το θέμα το οποίο εμεί έχουμε κοινοποιήσει και γνωστοποιήσει. Είναι κάτι το οποίο τίθεται σε ισχύ στο τέλος του διμήνου, εκτός αν τα δύο θεσμικά όργανα είναι κάτι διαφορετικό πριν από το δίμηνο αν δεν υπάρχει κάποια ένσταση για Στην αρχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι πρόκειται για μια κατοξιδότηση πράξη και θα πρέπει εμεί να δούμε πώ θα τεθεί σε ισχύ όσο γίνεται πιο σύντομα, γιατί αυτή η διαδικασία έχει διενεργοποιηθεί για την προετοιμασία αυτών των προγραμμάτων και ε, εταιρικών σχέσεων και για αυτό εμεί έχουμε επισήμω ζητήσει από το Κοινοβούλιο να αναλάβει τι σχετικέ ενέργειε, ούτω ώστε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτό τον στόχο της έγκυρης ενεργοποίησης και θέσης σε ισχύ. Thank you uh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κομισιόν. Τους εισηγητές τώρα θα ακούσουμε. Ξέχασα να σας πω ότι όταν λάβαμε το έγγραφο για να προετοιμάσουμε καλύτερα τη συζήτηση, η Γραμματεία χρησιμοποίησε τη γραπτή διαδικασία και σας πληροφόρησε ότι τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να θέσουν και επίσημα ερωτήματα ως αντιρρήσεις προς την κατεξουσιοδότηση πράξη. Δεν έχουμε όμως λάβει καμία τέτοια αντίρρηση. Λοιπόν, και τώρα πρώτα ο εισηγητής, ε, ποιος από τους δύο πρώτος, ε, δεν θέλετε πρώτα η κυρία, όχι, <coughs> όχι, ο Λαμπέρ. Εχθές Θελήσαμε να προετοιμάσουμε και εμείς τη συζήτηση. Αυτή η κατεξουσιοδότηση πράξη είναι η πρώτη από μια σειρά που θα πρέπει να εγκριθούν και σε αυτή την περίπτωση Υπάρχει το παρελθόν της, ε, υπήρξε ο τριμερής διάλογος, οι συζητήσεις υπό την Κυπριακή Προεδρία. Ήταν και ένα από τα πρώτα θέματα που συζητήσαμε τότε και συμφωνήσαμε το άρθρο 5 και το έγγραφο εργασίας της Κομισιόν Conduct now a να τα αναδιατυπώσουμε. Τώρα το βασικό είναι να δούμε το περιεχόμενο και να δούμε αν οι βασικές ιδέες έχουν ληφθεί υπόψη ε, στα διάφορα κεφάλαια, αν χρειάζονται αποσαφηνήσεις, αν υπάρχει επαρκής διαφάνεια για όλους τους εταίρους. Και το συμπέρασμά μας είναι ότι το κείμενο που έχουμε μπροστά μας συμφωνεί απόλυτα με ό,τι είχαμε συμφωνήσει καταρχάς ο, με βάση την αρχή της partnership. Ήδη ένα χρόνο πριν αν θυμάστε πόσο είχαμε χαρί γιατί τα κράτη-μέλη δέχτηκαν να συνεργαστούν στα πλαίσια του δεοντολογικού κώδικα που είχαμε συζητήσει το 2013. Τότε βέβαια δεν είχε ακόμη εγκριθεί αυτός ο κανονισμός, πάντων. Βλέποντας το περιεχόμενο χαιρόμαστε γιατί το κείμενο έχει αποσαφινιστεί, δεν χρειάζονται νομίζω προσθήκες και οι συνάδελφοι δεν εξέφρασαν καμία αντίρρηση σε αυτή τη διαδικασία. Είχαμε τη δυνατότητα επομένως να εφαρμόσουμε την μέθοδο της λεγόμενης έγκαιρης μη προειδοποίησης, μη αντίρρησης. Άρα αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις και εδώ μέσα, αν δεν ακουστούν τώρα ή και από άλλες επιτροπές αργότερα, μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία ταχείας μη αντίρρησης. Αργότερα σήμερα θα συνομιλήσουμε και με τον ίδιο τον Επίτροπο για τη δυνατότητα αυτή και θα δούμε τι θα γίνει. Νομικά πάντως Αυτά ισχύουν. Να ακούσουμε και άλλους αν έχουν τίποτα διαφορετικό να μας πούν. Η πρότασή μας πάντως είναι να δεχτούμε την διαδικασία αυτή ταχείας μη αντίρρησης ή πρόορης μη αντίρρησης. Δεν ξέρω αν έχει καμιά άλλη άποψη η Κομισιόν, αν να μας την πει. Αυτό πάντως θα έδειχνε σε όλους που όσους ασχολούνται με το θέμα ότι όλα αλήθηκαν υπόψη όπως έπρεπε. Δεν προτσέχασα τίποτε Κωνσταντζα. Όχι, αυτό ήθελα να σας πω. Και η πρόεδρος η κυρία Χιούμπνερ μπορεί να μας εξηγήσει τι ακριβώς θα είναι τα επόμενα βήματα. Ορίστε. Η Κωνσταντσα. Ο Λάμπερτ δεν ξέχασε τίποτα. Αλλά επί τη ευκαιρία μια που βλέπω πολλούς συναδέλφους σήμερα για πρώτη φορά το νέο έτος να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία και επιτυχίες και ευτυχία και βεβαίως έχουμε και τις ευρωεκλογέ φέτος και η δουλειά που έχουμε μπροστά μας ανεξαρτήτως ε, κόμματος νομίζω είναι καλό επιχείρημα για να πάμε στις ε, εκλογές και να το παρουσιάσουμε και νομίζω πως η γρήγορη υιοθέτηση των ε, εταιρικών αυτών σχέσεων πράγματι είναι κάτι το πολύ θετικό με τον Λάμπερτ. Ευχαριστώ να δώσω τον λόγο στους κοιόδες συζητητές, εάν θέλουν να πούν κάτι. Ναι. Η Ελίζα ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για την ιδέα που είχατε για την διαδικασία να διεξαχθεί όπως έγινε από τη γραμματεία. Πράγματι είχαμε αρκετό χρόνο να τα δούμε, να συζητήσουμε με τους συναδέλφους, να υπάρξει κάποια αντίδραση. Το συζητάμε στην Επιτροπή και μετά στην ε, ομάδα. Νομίζω πως ε, υπό τις συνθήκες αυτές, τις προεκλογικές, όπου τρέχουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα, είναι λογική αυτή η διαδικασία και μπορούμε έτσι να προετοιμαστούμε και να έχουμε και μια σαφή θέση αλλά η θέση νομίζω της ομάδας είναι πλέον σαφής και όταν ε, πηγαίνει και κάτι στη γραμματεία μπορεί να ελεγχθεί γι' αυτό θεωρώ πως ε, πράγματι είναι πάρα πολύ αποτελεσματική διαδικασία να το ξαναπώ δεύτερο για την Κομισιόν πολύ καλή εφαρμογή των όσων είπαμε. Είχαμε διαπραγματευτεί καιρό και η παρουσία της Κομισιόν έδειξε πως πραγματικά αντιλήφθηκε το νόημα των διαφόρων κειμένων και τα εφάρμοσε τέλεια κατά την άποψή μου. Και το επαληθεύσαμε όλοι. Ξέρουμε πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα για να είναι ισορροπημένο το κείμενο και πραγματικά θα χαιρόμουν να εγκριθεί και γρήγορα στο Συμβούλιο. Δεν ξέρω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα από πλευράς κομισιών. Γιατί ξέρουμε και την νομική κατάσταση, τις λεπτομέρειες του κανονισμού. Παρόλα αυτά καλό είναι τα κράτη-μέλη να γνωρίζουν επίσης πώς έχουν οι λεπτομέρειες του κώδικα συμπεριφοράς και να το έχουν γρήγορα και να το λάβουν βεβαίως και οι ενδιαφερόμενοι εταίροι για να ξέρουν ποιοι είναι οι κανόνες που πρέπει να τηρήσουν. Γι' αυτό καλό θα ήταν να εγκριθεί γρήγορα και κάτι ακόμα όταν εγκριθεί από το Συμβούλιο νομίζω καλό είναι η Κομισιόν να χρησιμοποιήσει τα δικά της μέσα για τη δημοσιότητα και για την εκπαίδευση των εταίρων γιατί η εμπειρία που είχαμε με αυτά τα οποία λέει ο κανονισμός και το τι είναι τα προγράμματα είναι πως ε, η κατάσταση των επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι αυτή που ήταν πριν από μισό χρόνο. Ε, αυτό θεωρεί το Συμβούλιο και δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλες διαφορές γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό στις πράξεις κατεξιοδότηση και σε αυτήν και στις επόμενες να δημοσιευτούν γρήγορα. Ο κώδικας αυτός συμπεριφοράς ρυθμίζει και τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και βεβαίω είναι ιδιαίτερα αγαπητός γι' αυτό προτείνω η Κομισιόν να κάνει μια καμπάνια δημοσιότητας προς ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται ε, ένα μεγάλο αριθμό οργανώσεων στα κράτη-μέλη αλλιώς θα μείνει μόνο ένα κομμάτι χαρτί. Πρέπει νομίζω να αποκτήσει ζωή, αλλά μπορεί νομίζω τώρα πραγματικά να προχωρήσει. Ευχαριστώ λοιπόν εδώ πέρα πάρα πολύ τους συμμετέχοντες. Jesus. Παναγία μου και Χριστέ μου, τι τις κάνατε. Δηλαδή, όταν είναι ε, χαρούμενη η Ελίζα Μπεθρέτερ, είμαι και εγώ χαρούμενη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος ε, σκιώδης ε, θέλει να μιλήσει. Πάμε στους επόμενους ομιλητές. Δεν βλέπω κανένα. Ο Ζικλάς είναι εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ε, συνεχίσω στη μητρική μου γλώσσα. Ναι, ναι, βάλτε τα ακουστικά. Ε, λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να Ας ευχαριστήσω την Κομισιόν και τον Λάμπερτ. Νομίζω πως ε, πράγματι απέδωσαν οι διαπραγματεύσεις ε, και το ζήτημα των εταιρικών σχέσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από τη χώρα μου, όπου έχουμε συζητήσει πολλές φορές το θέμα αυτό με τα συναρμόδια Υπουργεία και με την Κομισιόν, αλλά παρόλα αυτά δεν καταφέραμε να γνωρίζουμε την ε, οριστική ε, εκδοχή του κώδικα συμπεριφοράς. Οπότε καλό είναι να ε, τα γνωρίζουμε για να μπορέσουμε να το ψηφίσουμε το συντομότερο δυνατόν. Όσον αφορά δε την συχνή επικοινωνία. Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται μπορούν να συνεχιστούν τα πράγματα όσο έχουν γιατί δεν ενδιαφέρουν από την τελική εκδοχή άρα ελπίζω σε πάρα πολύ γρήγορη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τις ε, συμβάσεις αυτές και ε, δεν έχω και καμία αντίρρηση για τα όσα φαίνονται εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ. Γιάννη Ολμπρίχη. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τη γραμμή που προτείνουν και οι δύο εισηγητέ. Είναι μια σαφής και απλή διαδικασία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το ερώτημά μου απευθύνεται προς την Κομισιόν. Γιατί συζητάμε την ομοθεσία και, την και η πραγματικότητα βεβαίω είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Πόσο ξέρουμε, τέσσερα κράτη-μέλη ήδη έχουν στείλει την συμφωνία αυτή. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν ποια θα είναι η διαδικασία όταν εγκριθεί ο κώδικας συμπεριφοράς για τις συμφωνίες που έχουν ήδη αποσταλεί. Τι θα γίνει, θα πούμε πως ε, ότι έκαναν τα κράτη-μέλη, π.χ. η Πολωνία η οποία έστειλε τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης δεν συμφωνεί με τον κώδικα συμπεριφοράς, κατά το οποίο εγώ δεν ε, νομίζω ότι ισχύει. Ε, θα υπάρχουν λοιπόν δύο διαδικασίες, μία ex post και μία ex ante για αυτούς που είχαν στείλει. Το έγγραφο αυτό, ε, τι θα τους πούμε, δεν είναι σωστό και θα το στείλουμε πίσω. Είναι τεχνικό το ζήτημα, αλλά ε, θα πάμε στις χώρες μας και ο κόσμος μας ρωτάει τι γίνεται με, την με τη δικιά μας την ε, συμφωνία αυτή γιατί ο κώδικας συμπεριφοράς δεν είναι έτοιμος. Αυτό είπαμε και εμείς. Μετά τα το Συμβούλιο και είπαμε ήταν κώδικας διοντολογίας να, να θεσπίζεται, να υπάρχει και να τηρείται. Έχετε το λόγο. Θα σας προξενήσει έκπληξη αλλά και εμάς μας αρέσει αυτή η πράξη καταξιοδότηση γιατί βεβαίως συνήθως είμαστε πολύ αρνητικοί αλλά εδώ πέρα πραγματικά πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή περίπτωση μας εξέπληξε δύο ερωτήσεις έχω είναι βεβαίως ε, η γνωστή δυσπιστία που έχουμε για τους ε, αντιπροσωπευτικούς ε, εκπροσώπους και τις ε, οργανώσεις ομπρέλα ε, που λέτε. Τι, δηλαδή όποιος δεν ανήκει σε κάποια οργάνωση, η ομπρέλα, σε κάποια κλαδική οργάνωση δεν μπορεί να, να εκπροσωπηθεί. Είναι σημαντικό νομίζω αυτό. Επίσης ε, κάτι άλλο. Ποια οργανώσεις στον τομέα των μη διακρίσεων θα με ενδιέφερε. Αλλιώς ε, η διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και ο έλεγχος τους ε, σύμφωνα με τις αρχές αυτές αναφέρεται επίση, αλλά συνολικά νομίζω πως είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Δεν βρήκα κανένα σοβαρό παραθυράκι. Πολύ καλή δουλειά που κάνετε. Jens. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σήμερα νιώθω πάρα πολύ ικανοποιημένο και έχω να σα πω ότι από ό,τι γνωρίζω είσαι στην Σουηδία. αρχέ αρχές, κοινωνικοί εταίροι και αυτοί και αυτοί είναι ενθουσιασμένοι με τον κώδικα διοντολογία. Ξέρουν ότι έρχεται και τον περιμένουν. Το 2013 είχαμε επικρίσεις κατά τη κυβέρνηση γιατί δεν πριτάνευε στο έργο της κυβέρνηση στο πνεύμα αυτό και έχει ανοίξει ο μεγάλη κουβέντα στην χώρα μου. Οπότε και εμείς ενδιαφερόμαστε για το τι θα πει η Κομισιόν, τι θα πει στον, ε, στο, στο Γιάννη. Όμως, πάρα πολύ σωστά τα είπε ότι θα υπάρξει τεχνική αρρωγή τα είπε η Κομισιόν. Διότι επί 12 χρόνια συζητάμε το πώ θα χρησιμοποιήσουμε τεχνική αρρωγή, ούτω ώστε να μπορέσουμε ε, ε, τι οργανώσει ε, αυτέ να τι βοηθήσουμε. Πάει αυτή η χρηματοδότηση στις κρατικέ αρχές, χρηματοδοτεί το έργο τους σε αυτές τις διαχειριστικές αρχές, οπότε και εμείς θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουμε να δυναμώσουν την εταιρική αυτή σχέση. Επομένως, θα πρέπει και στο Συμβούλιο να πατήσουν γκάζι και να είναι ταχεία διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτή τη γενικότερη ατμόσφαιρα ειδονισμού που βλέπω θα ήθελα να σας πω ότι είναι πράγματι καλό το έγγραφο θα ήταν ακόμη καλύτερο αν εκ των προτέρων γραπτή διαδικασία είχαμε μερικές λεπτομέρειες για να δούμε μήπως χρειάζεται καμία βελτίωση. Πάντως είναι καλό έγγραφο. Δεύτερον, έχω δύο ανησυχιούλες. Πρώτον, γιατί δεν αναφέρεται ρητά ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών ενδιαφερομένων, μόνο οι σημαντικότεροι αναφέρονται και δεύτερον δεν αναφέρεται η δυνατότητα η τεχνική αρρωγή, το πρόγραμμα τεχνικής αρρωγής να ε, δημιουργήσει εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα για εκείνους που θα το αναλάβουν. Συζήτησα με τον Λάμπερτ, είναι βασικό τουλάχιστον σε μερικά κράτη-μέλη να δημιουργηθούν τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα, να δημιουργηθεί ένα είδος δομής, κάποια δομή εμπειρογνωμόνων εκτός πολιτικής επιρροής, τεχνοκράτες δηλαδή, κάτι σαν ευρωπαϊκή διοίκηση θα έλεγα εγώ, για να εκπαιδευτούν και οι περιφέρειες και τα κράτη-μέλη ώστε με έξυπνο τρόπο, όχι όπως να είναι, με έξυπνο τρόπο, με αποτελεσματικό τρόπο να μάθουν ποια είναι τα ωφέλη της πολιτικής συνοχής. Θα στείλω και επιστολή στον Πίτερ Μπρέγκοβιτς και θα την ξαναστείλω και στον κύριο Μπόισμαν, στον διευθυντή που είναι αρμόδιος για αυτά, διότι γενικά Γίνεται μεν, αλλά θέλω να μάθω αν αφού καθοριστούν τέτοια εθνικά προγράμματα εκπαίδευσης με εξαμηνιές εξετάσεις κλπ. και με την υποχρέωση των εκπαιδευτών να αποδείξουν να είναι ότι μπορούν να κάνουν κάτι στα κράτη-μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο λέει ότι θα οικοδομήσει διοικητικές ικανότητες σε μερικά κράτη-μέλη όπως και στη Ρωμανία, Ρουμανία, αλλά πρόκειται και για την κοινωνικοποίηση εδώ. Δηλαδή να υπάρξει πραγματική θετική επίπτωση, αποτέλεσμα να ε, αλλάξει θετικά η καθημερινή ζωή των πολιτών έτσι ώστε οι διοικητικοί όσοι εργάζονται στα δημαρχία κλπ να αλλάξουν συμπεριφορά. Και θα ήμουν και εγώ ακόμη ευτυχέστερος από ότι όλοι οι υπόλοιποι αν η Κομισιόν μας έδινε το πράσινο φως για ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ευχαριστούμε Βίκτορα. Πριν δώσω το λόγο. Πώς θέλεις και εσύ Α, όχι, δεν Έχω ακόμη μια πληροφορία και μετά θα ζητήσω από τον Νικόλαο της Κομισιόν να προσθέσει κάτι. Λοιπόν, δεν λάβαμε από καμία επιτροπή κανένα σχόλιο μέχρι τώρα. Λάβαμε όμως τρία σχόλια από τη γραμματεία. Τη γραμματεία. Με τρία θέματα τα οποία, για τα οποία συνεννοηθήκαμε με τους συνεισηγητάς. Ζητήσαμε και γνωμοδότηση από τη νομική μας υπηρεσία για αυτά τα τρία σχόλια για να δούμε αν θεσμοθετείτε καμία αντίρρηση και από ό,τι κατάλαβα από τη νομική υπηρεσία δεν υπάρχει νομικά λόγος να θέσουμε αυτά τα τρία προβλήματα ως σημαντικά προβλήματα. Ερωτώ λοιπόν τον Νίκολας Για πέστε μας τι φρονεί και η Κομισιόν για αυτά τα τρία σχόλια της Γραμματείας. Ζητήσαμε από τους συνεισηγητές και δύο άλλους συναδέλφους δεν ήρθαν όμως να μας δούνε άρα θα μας απαντήσει η Κομισιόν στο πρόσωπο του Νικολάου. Uh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ναι, να απαντήσω σε ερωτήσεις που ακούστηκαν. Να ξεκινήσω με το θέμα των ε, οργανώσεων, ομπρέλε και τον κίνδυνο που υπάρχει να μην εκπροσωπούνται οι μικρές οργανώσεις. Ε, πρέπει να δούμε τη διατύπωση, γιατί νομίζω πως ξεκαθαρίζει την πρόθεση. Όπως είπα, είναι πολύ σημαντικό στο της συμφωνίας που είναι στο εθνικό επίπεδο και βεβαίω για να υπάρχει μια αποτελεσματική συμφωνία πρέπει να έχουμε περιορισμένους αριθμούς, δεν μπορεί να έχουμε 300 εταίρους. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε μια αντιπροσωπευτικότητα. Αυτό το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 3.2 ε, είναι ε, ότι θέλουμε να διευκολύνουμε την συμμετοχή ε, και νομίζω αυτό διευρύνεται αν υπάρχει μία οργάνωση γενικότερη. Αλλά βεβαίως βλέπετε με τα παραδείγματα των συνδικάτων πως μπορεί να υπάρχει μια συνομοσπονδία συνδικάτων σε εθνικό επίπεδο που είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε μια οργάνωση ομπρέλα και έτσι μέσω ε, αυτής ε, της ε, οργάνωσης υπάρχει εκπροσώπηση για πολλά ξεχωριστά συνδικάτα. Το ίδιο και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Μπορεί να υπάρχει μία ένωση οτά έτσι ώστε να υπάρχει μία αντιπροσωπευτικότητα. Οπότε απλά αποσαφηνίζουμε το τι θα γινόταν ε, ούτως ή άλλως. Ε, απλά φροντίζουμε να εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα αντί να κάνουμε μια επιλογή κάτι που θα σήμαινε πως κάποιοι εκπροσωπούνται και κάποιοι άλλοι όχι. Όσον αφορά λοιπόν αυτά τα οποία μας είπε η γραμματεία από την Επιτροπή Απασχόλησης. Προσπάθησα να το πω στην εισαγωγή μου, γιατί δεν ορίζουμε εμείς εδώ πέρα το τι είναι ε, ένας τέτοιος οργανισμός ομπρέλα. Ε, εισάγεται μία έννοια και νομίζω είναι σαφές όταν ένας από τους εταίρους ε, έχει συστήσει έναν οργανισμό για να, ομαδοποιούν τα, για να ομαδοποιήσει τα συμφέροντά τους αλλά νομίζω η έννοια είναι σαφής. Ε, δεν είναι κάτι το νομικά περιοριστικό. Ελπίζω δηλαδή να μην θεωρηθεί πρόβλημα. Γι' αυτό το οποίο είπε τώρα ο Γιάνν Όλμπριχτ. Επανερχόμαστε σε ένα από τα ευαίσθητα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις. Τα κράτη-μέλη ανησυχούσαν να μην υπάρχει κάτι το αναδρομικό, γιατί ορισμού ο κώδικας συμπεριφοράς θα τεθεί ενισχύ μετά το βασικό νομοθέτημα, αλλά νομίζω πως εδώ τα κράτη-μέλη απαιτείται ούτως ή άλλως, σύμφωνα με το άρθρο 5, να σέβονται την αρχή αυτή. Άρθρο 40 παράγραφος 2 αναφέρει πως η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης πρέπει να προετοιμαστεί σε συνεργασία με τους εταίρους στο άρθρο 5. Η πρόεδρος αναφέρθηκε στην δήλωση που έγινε για να υπάρξει μια κατεύθυνση ότι δηλαδή τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν κάτι όσον αφορά και να δώσουν τους στόχους όταν ε, υπογραφεί η συμφωνία και το CPR το άρθρο 14 λέει πως τα κράτη-μέλη θα δίνουν πληροφορίες για το πως έγινε σεβαστή αυτή η αρχή της εταιρικής σχέσης. Η δε πράξη κατεξιοδότηση ε, λέει σε πιο μεγάλο βαθμό λεπτομέρεια... το ποια πρέπει να είναι αυτή η αρχή γιατί ορισμού όταν θα τεθεί ενισχύ Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υιοθετήσει ακόμα, δεν έχουμε εγκρίνει καμία τέτοια συμφωνία. Οπότε οι πληροφορίε που αναφέρονται εδώ πέρα αναμένουμε να περιέχονται σε κάποια τέτοια συμφωνία εταιρική σχέση και το αναμένουμε αυτό. Οπότε οπωσδήποτε δεν μπορούμε κατά να επιμείνουμε να μπουν κάποια στοιχεία του κώδικα συμπεριφοράς που αφορούν το παρελθόν, αλλά νομίζουμε πως δεν ε, θα υπάρξουν αντιφάσεις. Δεν θεωρούμε πως υπάρχει κάποιο κενό. Υπάρχει μια βάση νομίζω ε, για να θεωρήσουμε πως έχει γίνει σεβαστό το άρθρο 14 όσον αφορά την ε, συμφωνία με τους εταίρους και για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται νομίζω πως είναι επαρκής η βάση, δεν είναι τίποτα το προβληματικό στην πράξη και θα σεβαστούμε πλήρως τα όσα αναφέρονται στον κανονισμό κοινών διατάξεων και στην δήλωση όσον αφορά την μη αναδρομικότητα. Θα ορίσουμε το όριο σε ένα σημείο το οποίο ε, δεν θα είναι εφαρμόσιμο γιατί βεβαίως ο κώδικας συμπεριφοράς θα τεθεί ενισχύ τις επόμενες εβδομάδες. Για το θέμα των πληροφοριών συμφωνούμε πως πράγματι πρέπει η Κομισιόν να φροντίσει να υπάρχει ενημέρωση. Το έχουμε κάνει αυτό με τις προσπάθειες ε, που καταβάλαμε από όταν εγκρίθηκε η πράξη κατά εξουσιοδότηση και σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διατάξεις αυτές για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι αποτελεσματικό και οπωσδήποτε θα μπει αυτό στη διαδικασία παρακολούθησης ε, στην εφαρμογή του προγράμματος. Θα συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να είναι αποτελεσματικές αυτές οι επιτροπές ε, και ε, θα φροντίσουμε να γίνει σεβαστή πρόγραμμα η δέσμευση αυτή. Δεν θα είναι μόνο ένα κομμάτι χαρτί, θα πρέπει να έχουμε αποτελέσματα γιατί θα επανέλθουμε στην αξία μιας αποτελεσματικής εταιρικής σχέσης για ποιοτικά προγράμματα. Μετά είχαμε το άλλο θέμα της σχέσης με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είχαμε ένα ζήτημα ορολογίας τι σημαίνει άμεσα εμπλεκόμενη στα προγράμματα καθώς το άρθρο 7.4 ε, διαφέρει από το άρθρο 6.3 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αλλά δεν θεωρούμε πως αυτό έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία και οπωσδήποτε δεν είχαμε σκοπό την διαφοροποίηση από τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 6.3. Μιλάμε εδώ πέρα για τα προγράμματα αυτά. Σκοπεύουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τους κοινωνικούς εταίρους και τις ΜΚΟ ε, όταν ε, βεβαίω ε, τεκμηριωθεί η ανάγκη. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιος περιορισμός που προκύπτει από τη διατύπωση αυτή του άρθρου 17 παράγραφος 4. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε τώρα πρέπει μόνο να συμφωνήσουμε στα πορταθέντα. Έχει κανείς αντίρρηση με την διαδικασία μη αντίρρησης. Ε, Λαμπέρτο ρώτησα αν είναι κάποιος αντίθετος. Κανείς. Οπότε μπορώ να απευθύνω μία επιστολή προς την διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών να σας πω ότι μπορεί να συμβεί μέχρι την ε, εκπνοή της ε, προθεσμίας. Θα απευθύνω μία επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής των Πρόεδρων Επιτροπών. Ο κύριος Λένε θα ενημερώσει τους υπόλοιπους πρόεδρους. Οποιαδήποτε επιτροπή μπορεί να απορρίψει την ε, πράξη αυτή, όχι μόνο η Επιτροπή Απασχόλησης και αν δεν υπάρξει κάποια αντίρρηση εκεί θα πάει στην Ολομέλεια. Και βεβαίως εκεί πέρα κανονικά οι πολιτικές ομάδες έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν την άποψή τους. Οπότε σας τα λέω, ενημερώστε τους γνωστούς σας ε, ή κάποιον πρόεδρο επιτροπής που θα μπορούσε να έχει αντίρρηση. Πείστε τους να μην το κάνουν. Τελειώσαμε λοιπόν. Και θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το οποίο είπαν πολλοί, το ότι δεχόμαστε αυτή τη διαδικασία τώρα δεν σημαίνει πως και στο μέλλον θα γίνουν τα ίδια. Θα το δούμε κατά περίπτωση και οπωσδήποτε η επόμενη είναι πολύ πιο πολύπλοκη οπότε δεν θα ακολουθηθεί μάλλον η ίδια διαδικασία. Ναι, Λαμπέρ. Σας ευχαριστώ όλους για την γρήγορη υιοθέτηση του θέματος. Στην προηγούμενη συνάντηση είχαμε πει αυτό το οποίο είπε και ο Γιάνν Άλμπρεχτ, δηλαδή το τι συμβαίνει όντως στην κάθε χώρα. Ε, είναι κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό θέλουμε λοιπόν να φέρουμε τον κώδικα συμπεριφοράς κοντά στα έγγραφα που υπογράφονται και είχαμε την ιδέα μήπως γίνει μια επίσημη ακρόαση της Επιτροπής μας για να υπάρχει δυνατότητα να ακούσουμε τους ε, συμμετέχοντες εδώ πέρα. Νομίζω σημαντικό είναι να το συζητήσουμε αυτό και το απόγευμα. Τα είπε και ο κύριος Χάν. Τώρα έχουμε δηλαδή τον κώδικα συμπεριφοράς ε, και... Έτσι. Εντάξει, κάτι να κάνουμε όμως. Έτσι. Έτσι, ας σκεφτούμε λίγο πώς γίνει καμία κρόαση τις επόμενες μήνες. It's decided, I understood that we have agreed on this and decided, but... Uh, ναι, πράγματι, και εγώ χαίρομαι που συμφωνήσαμε και αποφασίσαμε. Λοιπόν, πώς να αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Περνάμε στο σημείο 6. Η ψηφοφορία της ε, Στέρας Φέγκουτ. Ε, είναι όμως 11 παρά 1. Έτσι. Ας περιμένουμε μήπως και μην και τυχόν. Uh, once Lambert takes his seat. Μόλις, μόλις καθίσει ο Λαμπέρ θα ψηφίσουμε. Πρώτα για το Ταμείο Αλληλεγγύης. We make this fake vote. What, what, what?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 Ο υπεύθυνο τη γραμματεία μα παρά την πενταετή του εμπειρία δεν ξέρει τι να μα συμβουλεύσει. Λοιπόν, τέλο πάντων, αρχίζουμε. Yeah, you Με τη συμβιβαστική πένδε ηλεκτρονικά. Υπέρ. Εκάτα. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Υπέρ. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ επαλήθευση για την 57 άρχη του ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 54 υπέρ Επαλήθευση και για την 54 άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Που δεν αποτέλεσμα. Ξανά. Γιατί το αποτέλεσμα εξαφανίστηκε. Την 54 ξανά ηλεκτρονικά. 54. έληξε απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 7 υπέρ αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται αιτιολογική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά εγκρίνεται, συμβιβαστική 1 υπέρ κατά εγκρίνεται, 21 υπέρ, επαλήθευση για την 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, 23 υπέρ, κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά εγκρίνεται. Α, όχι, κάποιο λάθος έχω κάνει. Κάποιο λάθος. 34 και 35 θεωρεί η κυρία Μπαράτσου ότι καλύπτονται, δεν τις ψηφίζουμε λοιπόν και περνάμε τώρα στη 37 ηλεκτρονικά. The vote is closed. Έληξε. Απορρίπτεται 36 υπέρ. 36 υπέρ είπα. Κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα από την Επιτροπή Προϋπολογισμών θα ψηφίσουμε μόνο την 8. Δεν έχετε μετάφραση προς τα Ιταλικά. Α, έχετε, εντάξει. Άντε, ψηφίζουμε λοιπόν την 8 της Επιτροπής Προπολογισμών. Υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Και 13 υπέρ, Κατά εγκρίνεται. Η τελική ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα χρειάζεται απλή πλειοψηφία ενώ για τις διαπραγματεύσεις 25 συν Να το ξέρετε λοιπόν. Για το νομοθετικό πρόταση. Πώς, πώς, πώς. Για την νομοθετική πρόταση άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικός. Έληξε εγκρίνεται 37 ψήφοι υπέρ 3 κατά και για το νομοθετικό ψήφισμα τώρα ηλεκτρονικά ε, άρχεται ε, ναι έλειξη εγκρίνεται και τώρα χρειαζόμαστε 25 συνέναν για την διαπραγματευτική εντολή και η διαπραγματευτική ομάδα θα είναι ο εισηγητής, η Σκιώδης και η πρόεδρος λοιπόν Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Έληξε. Υπάρχει, υπάρχει 38 ψήφοι Ευχαριστώ. Τελείωσε η ψηφοφορία αυτή. αυτή. Το έχω, ναι. Τώρα... Τώρα έχουμε την έκθεση της Αβυσάρ Τόμας όσον αφορά το, την 7η και 8η έκθεση πρόοδου και σας υπενθυμίζω ότι έχει αποσυρθεί η τροπολογία 22. Και, ο Θεέ μου, ξεκινάμε με την προφορική. Έχει κάνει ένσταση κατά της προφορικής. Αφορά αυτή τη διάταξη πριν την παραγράφω ένα από την έχουμε τώρα ε, αυτή είναι η προφορική υπέρ κατά εγκρίνεται και τώρα η συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πρόταση 14 απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 On amendment 13, the vote is open. 14. Ψηφίζουμε. Πέρας. 2 uh, in favor Συμβαστική 2 εγκρίνεται, συμβαστική 3 εγκρίνεται, απασχόλησης 13, ε, θα γίνει έλεγχος ηλεκτρονικός για την πρόταση 13 της Επιτροπής Απασχόλησης. Ψηφίζουμε τώρα. The vote is closed. Πέρασε και, και απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε την πρόταση 12. Έχει ε, απορριφθεί ε, τροπολογία 20 έχει. Εγκρίνεται. Έχει αποσυρθεί η 22 προφορική της εισηγητρίας. Ε, κάποιος κατά της προφορικής θα την ψηφίσουμε, τη εισηγήτριες προφορική υπέρ εγκρίνεται, συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, πρόταση. 4 γυναικών υπέρ κατά αποχές α, απορρίπτεται. Πρόταση 9 γυναικών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόταση 4 επασχόλησης υπερκατά. κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την πρόταση 4.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 Προφορική. Πριν την παραγραφό 9. Δεν υπάρχει ένσταση υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 29 υπέρ. 29 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 6α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική πριν την παραγραφό 11 υπέρ κατά. 11 δεν υπάρχει ένσταση υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 7 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 34 υπάρχει μια προφορική υπερκατά ποιος είναι κατά του 34 όπως έχει τροποποιηθεί έλεγχος για το 34 όπως τροποποιήθηκε από την προφορική Λαμπέρ, I, I do it for you because you were like... Λαμπέρ, για σένα το κάνω, γιατί σαν χέρι έδειχνες προς τα κάτω, τώρα έδειχνες προς τα πάνω. Ε, δεν θα, δεν θα πρέπει να σου κάνω τη χάρη. Close and it's nearly unanimously adopted. Σχεδόν ομόφωνη γίνεται. Πρόταση 2. Απασχόληση. Ποιοι είναι υπέρ. Απασχόληση υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να γίνει ένοχο για την πρόταση 2 της απασχόλησης. Δεν ξέρω το, το ΕΛΚ που το πάει. Ε, πρόταση 2 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Yeah, you just close the vote. And it is largely rejected. 35. Με ευρία πλειοψηφία απορρίπτεται. Against abstentions adopted. Amendment 38. 38 υπέρ. Κατά. Α, δεν ξέρω, γίνει έλεγχος για την τροπολογία 38. Ψηφίζουμε. Closed. Πέρας. Εγκρίνεται τροπολογία 40. Πώς? 40, 40. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Δεν ξέρω αν θα γίνει έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πρόταση 2 γυναικών υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πρόταση 3 γυναικών υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπερκατάποχε. εγκρίνεται πρόταση 6 γυναικών υπέρ κατά πρόταση 7 γυναικών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 γυναικών υπέρ αποχές εγκρίνεται 10 γυναικών υπερκατα κατά έλεγχος για το 10 The vote is closed. Πέρασε και απορρίπτεται. Αιτιολογικέ παράγραφοι έχουμε την τροπολογία παραθμών 1 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται δεύτερη τροπολογία υπέρ έλεγχος για τη δεύτερη τροπολογία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά έλεγχος για το 9. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική επί του 11. Κανείς δεν ενίσταται. Επόμενα ψηφίζουμε το 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πρόταση α γυναικών. Υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την πρόταση α γυναικών. Closed. Rejected. Και απορρίπτεται. Πρόταση β γυναικών. Α, ε, τώρα είστε κατά, υπέρ κατά, ε, απορρίπτεται. Οπότε πάμε για την ηλεκτρική ψηφοφορία, τελική ψηφοφορία υπέρ, κατά. Πέρας. 39 υπέρ, ένας κατά. Συγχαρητήρια. Vote on... Τώρα, περνάμε στην εκθέση Φρανσουά Αλφονσί. Νομίζω εδώ πέρα ο Λαμπέρ ε, κάτι θέλει να πει. Ναι. Εδώ πέρα η αρμοδιότητα της Επιτροπής μας είναι το αντικείμενο κάποιων ε, τροπολογιών που κατέθεσα και στην Ήτρε και εδώ πέρα. Όπως είδαμε σήμερα το πρωί, δεν είναι ακριβώς την αρμοδιότητά μας, αλλά θα ψηφιστούν στην, ε, κατά κύριο λόγο αρμόδια επιτροπή τα άρθρα 24, 12 και 14 ναι. και καταλήξαμε με τη γραμματεία πως δεν θα τα ψηφίσουμε εδώ πέρα γιατί ε, νομικά ανήκουν στους άλλους. Ε, αυτές είναι τροπολογίες, όχι άρθρα, λέει η πρόεδρος. 24, 12 και 14. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Καλύτερα να τα ψηφίσουμε, να ψηφιστούν στην Ήτρε ούτως ή άλλως. Ε, μου λένε πως είναι δική μου η αρμοδιότητα. Ωραία, συμφωνώ, όλος εξαιρετικός, λέει η Πρόεδρος. Χαίρομαι, λέει ο κ. Φανής, Ωραία, ξεκινάμε με τροπολογία 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 20 υπέρ. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 21 με 20. Γι' αυτό υπήρχε αμφιβολία. 21 υπέρ. Να την επαληθεύσουμε και αυτήν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 22 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 όχι, υπάρχει προφορική τροπολογία του Φρανσουά, είναι κανείς κατά, όχι, ωραία, την ψηφίζουμε. 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή, εκτιμώντας 1 υπέρ, να επαληθεύσουμε την τροπολογία 1, τον εκτιμώντας. Να έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 10 υπέρ. Μα την επαληθεύσουμε τη 10. Πέρας. 22 με 18. Εγκρίνεται. Ταυτόσημη, άρα δεν ψηφίζουμε. Δύο, λοιπόν. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε. Εγώ νομίζω ότι έχει περάσει, αλλά τέλος πάντων. Τροπολογία 2, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τέσσερα υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Έντεκα υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Απορρίπτεται. κατρία υπέρ. Κατά δεκτή. 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία Δεκτή, μάλιστα. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε, εγκρίνεται. Τώρα έκθεση Γκοτμάνης για τα στατιστικά στοιχεία. Τροπολογία 23 υπέρ. Να την επαληθεύσουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 24 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 25 υπέρ. Να την επαληθεύσουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές δεκτεί 27 υπέρ να επαληθεύσουμε την 27 πέρας απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές δεκτεί 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 υπέρ να επαληθεύσουμε 31 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Και δεκτή. 32 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 34, 5, 6, 37 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά 40 μέχρι 50 έχουν αποσυρθεί. Πάμε στα εκτιμώντας. 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8 και 9 είναι συμβατές ε, ψηφίζονται από κοινού. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτές. 10 υπέρ να την επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά αρχή τη ψηφοφορία. Πέρας. Τι κάναμε. Εντάξει, λάθος έκανα. Λοιπόν, δεκτή. Ε, πανερχόμαστε σε αυτή που νόμιζα ταυτόσημη, αλλά είναι συμβατή. 8 και 9 πρέπει να ψηφιστούν χωριστά. Λοιπόν, εκτιμώντας 3 τροπολογία 8 δηλαδή υπέρ να την δούμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Εννέα. Υπέρ. Βαλθεύουμε και την εννέα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Έντεκα. Υπέρ. Και αυτή θα την επαληθεύσουμε. Να έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 12, 13, 14 αποσύρονται. 15. Να την επαληθεύσουμε. Πέρας. 16 υπέρ. Ναι. Νομίζω το ίδιο είναι. Ε, οπότε εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 1 αποσύρεται 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 αποσύρεται 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3 αποσύρεται 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 καταπίπτει. 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την γνωμοδότηση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 39. Μία αποχή, μία ψήφος. Κατά συγχαρητήρια. Έχει έρθει ο Υπουργός. Σε δύο λεπτά θα είναι εδώ πέρα ο κύριος Χατζηδάκης, ο Υπουργός, Πρώην Ευρωβουλευτής, ο οποίος τώρα είναι προεδρεύων του Συμβουλίου, ελπίζουμε να έχει ήδη έρθει.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 Αρχίσουμε τη συνεδρίαση. Είναι η ώρα που έχουμε με την Προεδρία όπως δύο φορές το χρόνο. Και καλέσαμε τον Υπουργό Κωστή Χατζηδάκη που είναι και πρώην συνάδελφος πολλών από εσά εδώ στην Επιτρόπη μας. Remind also all of... Γι' αυτό σας υπενθυμίζω ότι θα συζητήσουμε την ε, ελληνική προεδρία σε σχέση με την ε, πολιτική συνοχής. Πρώτα θα μιλήσει ο Υπουργός και μετά θα γίνουν οι ερωταπαντήσεις. Thank you, President. I think it's ah, apparently oh, okay. better because of the cameras or fine, whatever. Fine, fine, okay. Thank you, President. Uh... Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, συνάδελφοι, αφού μαθημένος από τα παλιά. Λοιπόν, είμαι συγκινημένος, όχι μόνο επειδή ήμουν βουλευτής ε, για 13 χρόνια, από το 1994 μέχρι το 2007, αλλά και γιατί ήμουν πρόεδρος της ε, επιτροπής αυτής. Και στα... Όχι, ήμουν μέλος με συγχωρείτε της Επιτροπής και τα 13 αυτά χρόνια και άρα είμαι πολύ συγκινημένος ε, που είμαι εδώ πέρα σήμερα ως ε, Προεδρεύων του Συμβουλίου αλλά έχω μπερδευτεί κιόλα. δηλαδή εγώ εξακολουθώ να αισθάνομαι ευρωβουλευτής ακόμα και ειδικά μέλος ε, της Επιτροπής. Ε, δεν τα λέω έτσι αυτά για να σας κολακεύσω, πιστέψτε με, έτσι νιώθω. Τέλος πάντων. Πρέπει τώρα να αναφερθώ στις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας. Είναι πρόκληση για εμάς, διπλή πρόκληση θα έλεγα για τους Έλληνες, γιατί πρώτα απ' όλα η προεδρία αυτή συμπίπτει με τις ευρωεκλογές μια στιγμή προφανώς κρίσιμη. Πρέπει να κλείσουν ορισμένα θέματα και να στείλουμε κάποια θετικά μηνύματα και επιπλέον είναι και ευκαιρία για εμάς να επανορθώσουμε τη ζημιά που έχει γίνει στην εικόνα της χώρας τα τελευταία χρόνια. Οπότε θέλουμε να αρπάξουμε αυτή την ευκαιρία και να σας εκπλήξουμε θετικά, όχι με μια πολύ φιλόδοξη, πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Θαύματα δεν μπορούν να γίνουν σε έξι μήνες ή σε τρεις καλύτερα. Αν λάβουμε υπόψη και τις ευρωεκλογέ και το ότι το Κοινοβούλιο θα διαλυθεί στα μέσα του Απριλίου. Θα προσπαθήσουμε να σας ε, καταπλήξουμε μέσω αποτελεσμάτων με το να έχουμε κάποιες συγκεκριμένες προοπτικές και κάποια απτά αποτελέσματα τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου, σε συνεργασία πάντα με τα άλλα κράτη-μέλη, γιατί έχουμε την Προεδρία αλλά δεν έχουμε ψευδεστήσεις, ξέρουμε πως εμείς ε, μόνο το ρόλο του καταλήτη μπορούμε να παίξουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και πάντα σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Γιατί ε, συνεργαζόμαστε επίσης όρις. Τώρα η συναπόφαση δεν είναι πλέον η εξαίρεση όπως ήταν το 1994 όταν πρώτο ήρθα στο Κοινοβούλιο είναι ο κανόνας. Οπότε πρέπει να συνεργαστούμε με αμοιβαίο σεβασμό και κοινού στόχους. πολιτική συνοχής. Είναι οπωσδήποτε θεμέλιο λίθος τη Ευρώπη, ειδικά τώρα. Έτσι όπως πάει και η ύφεση στην Ευρώπη, τη στιγμή που προσπαθούν κάποια κράτη-μέλη να επιστρέψουν στην ανάπτυξη, η πολιτική συνοχής έχει μεγαλύτερη σημασία. Είναι το βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά για να αντιμετωπίσει την κρίση οικονομικά μιλώντας. Είναι ένα μέσο βασικό για να στηρίξει τους ε, κύριους στόχους της στρατηγικής ε, της Ευρώπης 2020 για να έχουμε ισορροπημένη και αποκεντρωμένη ανάπτυξη που θα προωθήσει την περιφερειακή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μειώσει τις ανισότητες. Υπό αυτές τις συνθήκες η Ευρώπη πρέπει να εστιαστεί σε μια συζήτηση για ένα φιλόδοξο και ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση σύμφωνα με τη στρατηγική 2020 για να δημιουργήσει και θέσεις εργασίας. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στην επιτυχία των διοργανικών διαπραγματεύσεων για το πακέτο συνοχής του 2014-2020 που οριστικοποιήθηκαν Επιληθανικής προεδρίας. Είχα την ε, τιμή και το προνόμιο και στο παρελθόν ε, το 1999 και το 2005 να λάβω μέρος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Εν πάση περιπτώσει και χωρίς την δική μου παρουσία ήταν επιτυχής οι διαπραγματεύσεις. Οπότε θα θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου για την επικοδομητική στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλη τη διαδικασία, ειδικά της ε, Προέδρου της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Πολιτικής, κυρία Χιούπνερ, ε, των εισηγητών και οπωσδήποτε των διαπραγματευτών. Η διακτήμηση βεβαίως απευθύνεται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπετε συνεργαζόμαστε και με την Κομισιόν Οπότε πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις μαζί τους. Είμαι σίγουρος πως ε, συμφωνείτε μαζί μου πως η επιτυχής ολοκλήρωση των διοργανικών διαπραγματεύσεων είναι ακόμη πιο ικανοποιητική καθώς ξέρουμε πως είναι η πρώτη φορά που είχαμε την τακτική νομοθετική διαδικασία της συναπόφαση που χρησιμοποιήθηκε για ολόκληρο το πακέτο της συνοχής. Σημαντικό αυτό για την Επιτροπή, σας ε, για το Κοινοβούλιο για την Ευρώπη. Ξέρετε πως, το ξέρετε καλύτερα από μένα, χρειάστηκαν πάνω από 100 συνεδριάσεις στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου για να έχουμε μια επιτυχή κατάληξη και σημαντική πολιτική ευελιξία από όλους τους εμπλεκόμενους. Μόνο χάρη σε αυτήν την ευρηματική και αποτελεσματική συνεργασία οριστικοποιήθηκε το πακέτο αυτό στο τέλος του 2013 και ετέθη ενισχύ εγκαίρος. Βεβαίως, αυτό ήταν η έγκριση του κανονισμού. Τώρα περνάμε στην επόμενη φάση. Λιγότερο δύσκολη πολιτικά, αλλά δεν ξέρω αν είναι λιγότερο δύσκολη από τεχνική σκοπιά. Έχουμε την εμπειρία, έχουμε πρώην επίτροπο εδώ και όλοι σας γνωρίζετε πως ο διάβολος όπως λένε κρύβεται στις λεπτομέρειες. τότε η Ελληνική Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε η εφαρμογή του πλαισίου του νομοθετικού πακέτου να είναι όσο δυνατόν πιο αποτελεσματική. Η απόφαση να έχουμε άτυπο συμβούλιο των Υπουργών που είναι αρμόδιοι για την ε, συνοχή τον Απρίλιο στην Αθήνα καταδεικνύει ε, τη σημασία που αποδίδουμε στην πολιτική αυτή όσον αφορά την καταπολέμηση της ύφεσης και της ανέργειας. Η Ελληνική Προεδρία ελπίζει ε, το άτυπο αυτό συμβούλιο να μην είναι απλά έτσι μια συζήτηση ακαδημαϊκή. Εντάξει, οι υπουργοί θα έχουν και άλλες ευκαιρίες να κάνουν ταξιδάκια στην Αθήνα και αλλού. Θέλουμε πραγματικά να δούμε σοβαρά το, τις διατάξεις των κρατών μελών που θα εφαρμόζουν τον νέο κανονισμό. Η συμβολή της Κομισιόν θα είναι κέρια καθώς θα δοθούν χρήσιμες κατευθύνσεις για την γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων. Το ζήτημα αυτό το συζήτησα ήδη με την κυρία Χιούμπνερ, την ε, προσκάλεσα να παραβρεθεί στην συνάντηση αυτή και αν θέλετε κι εσείς ευχαρίστως. Α, έχουμε χρόνο να τα οργανώσουμε αυτά. <coughs> Αλλά θέλουμε παρουσία του Κοινοβουλίου και εγώ προσωπικά θέλω για προφανείς λόγους. Όσον αφορά τώρα τις προκλήσεις ε, για το προσεχές μέλλον, το ζήτημα των πράξεων κατεξιοδότηση πρέπει επίσης να αναφερθεί. Παρά το ότι η διαδικασία λήψη αποφάσεων είναι παράλληλη στο Συμβούλιο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σαφές πως το θέμα αυτό θα απαιτήσει εκτεταμένες συζητήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Και πρέπει να είμαι ειλικρινής. Η Κομισιόν αποφάσισε να εκδώσει λίγες πράξεις κατευσιοδότηση με πολλά άρθρα. Έτσι πιθανώς να έχουμε καθυστέρηση της όλης διαδικασίας, καθώς κάποια κράτη-μέλη μπορούν, μπορεί να απορρίψουν ολόκληρο το πακέτο, γιατί μπορεί να έχουν μια αντίρρηση σε ένα ή πολλά στοιχεία του πακέτου. Ακόμα και ένα μόνο. Ήδη η Κομισιόν έχει δηλώσει έχει στείλει στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο τον κώδικα συμπεριφοράς και εμείς ε, σκοπεύουμε να πούμε εξ αρχής πως δεν έχουμε αντίρρηση έτσι ώστε να υιοθετηθεί στην επίσημη εφημερίδα πριν εκπνεύσει η δίμηνη περίοδος που προβλέπει η συνθήκη. Ενώπιση των ευρωεκλογών Θεωρώ πως πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα για το πόσο εκτιμούμε τον ρόλο των κοινωνικο-οικονομικών φορέων. Αλλά το ζήτημα αυτό των πράξεων κατεξοδότηση και το πώς θα το δούμε και στο επίπεδο του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου είναι προτεραιότητα για εμάς. Είναι τεχνικό ζήτημα, αλλά μπορεί τελικά να γίνει και θέλω να με μαζί σας πολιτικό ζήτημα. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε στενά με τα άλλα κράτη-μέλη, με το Κοινοβούλιο και με την ε, Κομισιόν, ειδικά με τον κύριο Χάν, για να μην έχουμε καθυστερήσεις για λόγους οι οποίοι δεν είναι σημαντικοί και είναι κρίμα να καθυστερήσει όλη η διαδικασία παρά το ότι θα έχουν εγκριθεί εγκαίρως οι κανονισμοί και θα είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε στους πολίτες. Γιατί καθυστερεί δηλαδή η εφαρμογή των νέων κανονισμών λόγω νομικών ζητημάτων. Τώρα, θα αναφερθώ σε ένα άλλο σημαντικό ζήτημα και χαίρομαι που είναι εδώ η συγκήτρια η κυρία Στέρας το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Θα ήθελα να πω πως η έγκριση του τροποποιημένου κανονισμού είναι οπωσδήποτε προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας. Και πώς αλλιώς. Οι διοργανικές διαπραγματεύσεις ε, υπό το στην απόφαση. πρέπει να ξεκινήσουν σύντομα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και να οριστικοποιηθούν με τρόπο αποτελεσματικό και γρήγορο το αργότερο τέλος Μαρτίου. Θεωρώ πως θα συμφωνήσετε όλοι στην συμφωνία των διαπραγματεύσεων καθώς ενώ σε γενικές γραμμές ανταποκρίνεται στους στόχους του το μέσο αυτό θεωρείται πως δεν μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς καθώς κάποια κριτήρια για την ενεργοποίησή του είναι πάρα πολύ πολύπλοκα ή δεν είναι αρκετά σαφή. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τροπημένο κανονισμό είναι μια σημαντική ευκαιρία για μεταρρύθμιση καθώς αδλούμε διδάγματα από την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής προτείνουμε λύσεις για να γίνει πιο απλό στην χρήση του ταμείου και να έχει σαφέστερα κριτήρια για το ποιος μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Τέλος, η πρόκληση δεν είναι μόνο η πίεση χρονική, που είναι το προφανές, αλλά, κυρία Εστέρας, έχουμε και τους περιορισμούς του προϋπολογισμού και δεν ομιλώ εδώ πέρα ως υπουργό Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά ως Προεδρεύον του Συμβουλίου. Καταλαβαίνετε τι ήθελα να πω και είμαι σίγουρος πως η συνεργασία της Επιτροπής σας με το Συμβούλιο θα συνεχιστεί και σκοπεύουμε να εγκριθεί αυτή η πρόταση πριν από τις ευρωεκλογέ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα, μπορούμε να στείλουμε στους πολίτες. Είναι κάτι κατανοητό από όλους. Είναι μια έκφραση απτή της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Οπότε θα ήταν κρίμα να μην καταλήξουμε σε μια συμφωνία, σε ένα κοινό παρανομαστή πριν από τις ευρωεκλογές για το θέμα αυτό. Και καταλήγω με τις εξόχως περιφερειακές περιοχές. Ε, καθώς προέρχομαι από μια χώρα νησιωτική αντιλαμβάνομαι πλήρως τις ιδιαιτερότητες των εξόχως περιφερειακών περιοχών. Οπότε, σας επιβεβαιώ πως η Προεδρία σκοπεύει να εγκρίνει όλα τα καθεστώτα που εκκρεμούν για τις περιοχές αυτές. Εκτιμούμε πάρα πολύ τη γνωμοδότηση της, ε, τη γνώμη της ε, Επιτροπής σας. Δεν υπάρχει εδώ πέρα διαδικασία απόφαση ε, αλλά ούτως ή άλλως εκτιμούμε την άποψή σας και πριν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τα ζητήματα αυτά αναμένουμε τις απόψεις σας. Οπότε είναι σαφείς οι προτεραιότητες μας. Πρώτα απ' όλα εφαρμογή του κανονισμού, των κανονισμών, δεν ε, εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από τα άλλα κρατημέλη και την Κομισιόν βεβαίω. Γι' αυτό θα έχουμε το άτυπο Συμβούλιο Συνοχής ε, τον Απρίλιο το οποίο θα το αφιερώσουμε μόνο σε αυτό το ζήτημα πώς θα επιλύσουμε τα προβλήματα στα κράτη-μέλη, πώς θα επιταχυνθεί η ανάπτυξη. Αυτό θέλουμε όχι να χάνουμε χρόνο. Δεύτερον, να δούμε τα τεχνικά και νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση και βεβαίω έχουμε τα δύο νομοθετικά πακέτα το Ταμείο Αλληλεγγύης που είναι σημαντικό και τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές που δεν είναι ζήτημα βεβαίως για κάποια καρατιμέλη αλλά για τις περιοχές αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχονται και ευρωεκλογέ, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά αυτό ούτως ή άλλως γιατί θέλουμε να αποδείξουμε πως οι Έλληνες μπορούν να έχουν αποτελέσματα, μπορεί να είναι επιτυχημένη η ελληνική προεδρία, γνωρίζουμε πως είμαστε καταδικασμένοι να επιτύχουμε και νομίζω θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Όπως γνωρίζετε από την προηγούμενη εμπειρία σας θα μιλήσουν οι συντονιστές και την Ο κύριος Βανίστελροι πρώτος. Ναι, έχουμε μια ώρα, θέλουν βέβαια πολλοί να μιλήσουν. Θα προσπαθήσω λοιπόν να συντομεύσω. Κύριε Κώστα Χατζηδάκη, σας ξέρουμε, ξέρουμε ότι έχετε πολύ γλυκιά προσωπικότητα, πολύ ευγενική, αλλά μπορείτε να είστε ελπίζω και σκληρός διαπραγματευτής. Και εμείς έτσι θα είμαστε, μην παρεξηγείτε. Αυτά τα θέματα για το Ταμείο Αλληλεγγύης, ας πούμε, θέλουν κάποια επιμονή. Συνήθως όλα αυτά απαιτούν κοινέ ευθύνες και συνεργασία. Λοιπόν. to say from Greece love. Oh, what Λοιπόν. Καλό είναι που το Συμβούλιο δείχνει την αποφασιστικότητά του και για τα διαρθρωτικά ταμεία ζητήθηκαν αλλαγέ και μερικέ χώρε είπαν ότι πρέπει να βελτιωθεί η πληροφόρηση των πολιτών, η επικοινωνία με τους πολίτες. Και εν ώψη και των εκλογών χρειάζεται κάποια θεματική συγκέντρωση, εξ συμφωνία. Ζητώ λοιπόν τη συνεργασία σας για να αναλάβουμε κοινέ δεσμεύσεις για καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών. In some country. Ξέρετε καλά πόσο σημαντικά είναι και στην Ελλάδα αυτά με την κρίση πόσο θα μπορούσαν να ωφελήσουν ας πούμε τις δημόσιες επενδύσεις και τις επιχειρήσεις um, αν υπάρξει καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία. Επενδύστε λοιπόν στην επικοινωνία και θα ήθελα να γίνετε εταίρος, συνεργάτης μας σε αυτό και για τις αλλαγές στις προοπτικές που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Χαίρομαι επίσης ιδιαίτερα που μιλήσατε και για την άποψή μας για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Look to your suggestion whether technically it can be taken on board. Φυσικά δεν πρόκειται εδώ για επιλεκτική προσέγγιση cherry picking αλλά και για το Ταμείο Αλληλεγγύης καλά μας τα είπατε. Θα μιλήσει και η κυρία Εστέρης βέβαια γι' αυτό. Αλλά εδώ και πολλά χρόνια, οπότε τότε που ήσασταν εσείς στο Κοινοβούλιο, επιμέναμε γι' αυτό το θέμα. Και ξέρετε πού πήγαν στραβά τα πράγματα. Στο Συμβούλιο πάντοτε στο Συμβούλιο ήταν ο κόμπος, δεν τελείωσε ποτέ η διαδικασία και ελπίζω να εφαρμόσετε όντως την δέσμευσή σας να γίνουν τα πράγματα πιο ελαστικά φυσικά. Υπάρχει η άτυπη συνάντηση που έχουμε και θα έχουμε, όπως γίνεται συνήθως. Το Κοινοβούλιο είναι διατεθειμένο να επιδείξει, να ενδιαφερθεί για τα πράγματα και για την ελληνική κατάσταση όπως έκανε και στο παρελθόν με την Task Force την πρόσκληση αυτή την παίρνουμε πολύ σοβαρά. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και αυτά είχα να σας πω. Κοιτάξτε. Η ε, για μισή ώρα ακόμα θα υπάρχει. Ε, στα υπόψη. Λοιπόν, Κωνσταντσε, ευχαριστώ Ντανούτα. Καλώς ήρθατε. Ξανά, Κώστα, στην Επιτροπή μας. Και οπωσδήποτε εύχομαι και σε εσά και στην Ελλάδα επιτυχημένη Προεδρία. Αυτό δεν βοηθάει μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να σταλεί το μήνυμα πώς ε, μπορείτε ως ε, μέλος Ένωσης να ασκήσετε μια επιτυχημένη προεδρία. Και βεβαίως, άκουσα τους στόχους σας, ε, οριστικοποιήσαμε νομίζω την βάση του πακέτου της μελλοντικής πολιτικής συνοχής δεν τα καταφέραμε όλα όσα θέλαμε, αλλά νομίζω τώρα έχουμε μια ε, καλή και σύγχρονη βάση για πολιτική συνοχή στα επόμενα 7 χρόνια. Τώρα πρέπει να δούμε τις ε, πράξεις ε, κατ' εξουσιοδότηση. Πράγματι, είπαμε να ξεκινήσουμε και την διαδικασία μη αντίρρησης για τον κώδικα συμπεριφοράς Οπότε στέλνουμε και εμείς το μήνυμα πως θέλουμε να επιταχυνθεί η οριστικοποίηση της ε, πολιτικής συνοχής. Και βεβαίως ελπίζουμε το μήνυμα να είναι σαφές προς το Συμβούλιο ότι εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να βοηθήσουμε τα πράγματα αλλά βεβαίως τώρα η Προεδρία, το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη πρέπει και αυτά να κάνουν ε, τη δουλειά τους. Δεν είναι, όπως είπατε, τεχνικό ζήτημα το να έχει κανείς ε, κάποια αμφιβολία. Ε, χρειάζεται και ένα πολιτικό μήνυμα πως ε, και τα κράτη-μέλη θέλουν να οριστικοποιηθεί το πακέτο αυτό της πολιτικής συνοχής. Κατόπιν Ταμείο Λεγγύης. Θα θυμάστε σίγουρα πως πριν από 7 χρόνια είχαμε την ίδια ακριβώς κατάσταση ότι δηλαδή έπρεπε να δουλέψουμε εμείς στο Κοινοβούλιο για ένα Ταμείο Συνοχής και το απέριπταν μετά επί σειρά ετών ε, τα κράτη-μέλη. Τώρα η κατάσταση είναι διαφορετική, είμαστε και στη συναπόφαση, αλλά εάν ε, επιτύχετε σε αυτό θα είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό γιατί 7 χρόνια απόρριψης από το Συμβούλιο και τώρα 3 μήνες διαλόγων και διαπραγματεύσεων. Αν τα καταφέρετε θα είναι φοβερό, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα νέο ταμείο αλληλεγγύης και νομίζω πως τώρα έχει φτάσει η στιγμή να τελειώσει κάποτε αυτή η υπόθεση και εύχομαι κάθε επιτυχία και νομίζω πως οι συγητής και οι σκιώδεις συγητές ε, είχαν δεσμευτεί και σκοπεύουν να έχουμε μια επιτυχή κατάληξη μέχρι το τέλος ε, της θητείας. Ευχαριστώ Ιβας Γκουτμάνης για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και εγώ θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Ξέρετε πως έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο στο Κοινοβούλιο. Μην περιμένετε λοιπόν ε, φοβερή δραστηριότητα, οπότε η δική σας ευθύνη είναι ακόμη μεγαλύτερη. Κάποια πράγματα ήθελα να αναφέρω. Κάθε περίοδος ξεκίνησε με διαφορετικές συνθήκες. Πριν 2007 ε, μέχρι τώρα είχαμε ξεκινήσει με τα διαφορετικά διαχειριστικά συστήματα και εκεί πέρα ε, βεβαίως είχαμε και το πρόβλημα εκεί πέρα οφείλονταν η καθυστέρηση εδώ πέρα λοιπόν τώρα έχουμε ακριβώς ε, το θέμα των συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου μόνο τρεις ή το πολύ τέσσερις χώρες έχουν στείλει στην ε, Κομισιόν την ε, συμφωνία. Ε, πάρα πολύ μικρό αριθμό γιατί υπήρχε ο χρόνο να προετοιμαστούν τα κράτη-μέλη για τι συμφωνίε αυτέ. και κάποιο πρέπει να δει το γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει γρήγορα. Το τρίτο θέμα που ήθελα να αναφέρω είναι το πρόβλημα με την ανεργία των νέων. Ε, η χρηματοδότηση είναι η πιο πολύ στην αρχή. Έχει μεγάλη σημασία βεβαίως ποια είναι η ποιότητα των προγραμμάτων. Μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Δεν είναι ένα κλασικό πρόγραμμα γιατί δεν υπάρχει κάτι τέτοιο εντό συνοχή. Υπάρχουν ε, προτεραιότητες με 11 σημεία, ε, ποσοτικούς δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν, αλλιώς ε, δεν θα πληρωθεί ένα ποσοστό. Και εγώ θα χαιρόμουν να δώσετε βάρος εδώ πέρα για το πώς ξεκινά αυτά τα προγράμματα κομισιών και πώς σε τελική ανάλυση θα έχουμε κάποια αποτελέσματα. Τέλος για την Ελλάδα. όχι μόνο όμως. Κάτι ε, δεν πάει καλά με το κοινωνικό ταμείο. Γιατί αν δείτε τις προβληματικές ε, χώρες, ε, μιλάω μακροοικονομικά προβληματικές, η Ελλάδα πολύ καλή στην Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, και Ταμείο Συνοχής είστε στην πέμπτη θέση το 2007-2013 72% απορρόφηση 10% πάνω από το μέσο όρο καλύτερη από την Ισπανία που επίσης δεν τα πάει άσχημα και καλύτερη από την Πορτογαλία που είναι ε, και αυτή αρκετά καλά. Αλλά αν δει κανεί το κοινωνικό ταμείο που σχετίζεται με την ε, ανεργία και τα υπόλοιπα, τότε η κατάσταση εκεί είναι διαφορετική. Είστε κάτω από το μέσο όρο. Είστε 15η χώρα στις 27 μαζί με την Ισπανία και είναι ενδιαφέρον οι χώρες οι οποίες έχουν την υψηλότερη ανεργία έχουν χαμηλή απορρόφηση του κοινωνικού ταμείου. Ίσως ένας λόγος είναι πως δεν υπάρχει εποπτεία της εφαρμογής. Όταν αρχίσαμε να υποβάλουμε προτάσεις ε, για το ποιος θα είναι υπεύθυνο για την εποπτεία του Ταμείου Συνοχής, εγώ υπέβαλα μία πρόταση, αλλά έπρεπε να την αποσύρω γιατί υπήρχε ζήλια. Κανείς δεν ήθελε να είναι αρμόδιος, ούτε η Ρέτζη, ούτε η Επιτροπή Απασχόλησης, ε, ούτε κανείς. Οπότε, ποιος είναι υπεύθυνο. Τελικά πέρασε μισός χρόνος. Γιατί πρέπει να δούμε πώς θα αναλύσουμε αυτά τα νούμερα. Αλλιώς θα μας κατηγορήσουν. θα μας κατηγορήσουν ότι δεν ξοδεύουμε τα λεφτά οι εχθροί της συνοχής. Μας λένε όλα λεφτά θέλετε και δεν τα κάνετε κάτι. Ξέρετε μέχρι τώρα έχουμε μέση απορρόφηση 64% και ε, στο κοινωνικό ταμείο και 60% στο ταμείο συνοχής κτλ. Αλλά 52% στις χώρες που τα πάνε χειρότερα στην συνοχή και στο περιφερειακό και ε, αυτές οι χώρες είναι και κάτω από τον μέσο όρο της απορρόφησης. Ε, θα πρέπει λοιπόν να ρίξετε βάρος στο κοινωνικό ταμείο και στην στο θέμα της ενέργειας των νέων. Ότζι Βλάσσακ, να ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις πρώτα. Και, και εγώ σας καλωσορίζω, Κωστή. Είναι μεγάλη χαρά για μας η παρουσία σας. Λοιπόν, πρώτον, θα ήθελα να τονίσετε περισσότερο ότι η πολιτική συνοχής είναι από τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας για την καταπολέμηση της ύφεση και της ανεργίας. Αλλά επίσης μια άλλη προτεραιότητα που είναι πολύ σημαντική την στήριξη της ανταγωνιστικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας. Ξέρουμε τα προγράμματα COSME και ορίζον και πρέπει να υπάρξει άμεση στήριξη των επενδύσεων. Έχετε καμία καινούρια ιδέα πώς να βελτιωθούν τα πράγματα εκεί. Τέλος, τέλος το διοικητικό άχθος. Αυτό είναι ο εφιάλτης μας. Αυτό. Έχετε καμία καινούργια ιδέα περί αυτού, μπορείτε να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε τα πράγματα και γι' αυτό. Κύριος Αγκουράκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αντιλαϊκή πολιτική και τα αντιεργατικά μέτρα εφαρμόζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξάρτητα αν οι χώρες βρίσκονται σε μνημόνιο ή έχουν μεγάλα ελλείμματα ανεξάρτητα αν έχουν χαμηλούς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτά τα μέτρα εφαρμόζονται σε βάρος των εργαζομένων, σε βάρος των μισθών και των κοινωνικών τους κατακτήσεων, γιατί το μεγάλο κεφάλαιο και τα μονοπόλια θεωρούν ότι μόνον έτσι μπορούν να βγουν από την κρίση που μαστίζει αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση, διατηρώντας και αυξάνοντας ταυτόχρονα την κερδοφορία του κεφαλαίου. Παρ' όλα αυτά ξέρετε ότι η ύφεση συνεχίζει να υπάρχει, οι προοπτικές για την ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερές και όσον αφορά ε, τα ζητήματα που ε, διαπραγματεύεται η πολιτική συνοχής, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερο, ακριβώς γιατί η οικονομική κρίση θα οξύνει τον ανταγωνισμό και θα οξύνει την ε, ανισόμετρη ανάπτυξη των διαφόρων κρατών και των περιφερειών. Ε, θέλω να ξέρετε όσον αφορά την Ελλάδα παραδείγματο χάρη, αυτό είναι και ο λόγο ακριβώ, αυτή η συνολικότερη πολιτική που έχουμε αλλαγή στο περιεχόμενο τη πολιτική συνοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι η πολιτική συνοχή καλείται να εξυπηρετήσει του στόχου τη Ευρώπη 2020 που ακόμα περισσότερο εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών και των τεχνολογικά προηγμένων ε, επιχειρήσεων με παράλληλη ε, ε, επιβολή νέων αντεργατικών μέτρων γιατί όπως σημειώνονται και στα εξάμεινα και ξέρετε ότι αυτά είναι υποχρεωτικά για τις όλες χώρε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ανταγωνιστική σε σχέση με την Ινδία και την Κίνα με αντίστοιχους μισθούς. Αυτή είναι η βασική κατεύθυνση, ε, σε αυτή την πορεία πορεύεται, γι' αυτό και όλα και η πολιτική συνοχή αυτού του στόχου θα εξυπηρετήσει και όχι τι αυξανόμενε φυσικά ε, κοινωνικέ και ε, λαϊκέ ανάγκε, γιατί κανεί δεν μπορεί να σταματήσει την εξέλιξη. Τα πράγματα γίνονται ιδιαίτερα δραματικά στην Ελλάδα που θέλω να ξέρουν οι συνάδελφοι ότι έχει υπολογιστεί ότι η μεγάλη ανεργία που έχει η χώρα μου, 27% και 62% στους νέους, θα μειωθεί στο μισό στα επόμενα 20 χρόνια εάν η Ελλάδα εξασφαλίσει έναν ρυθμό ανάπτυξης του 5% το χρόνο. 5% το χρόνο χρειάζεται η Ελλάδα για να μειώσει στο μισό την ανεργία που την ε, ε ταλανίζει τώρα. καταλαβαίνετε κανένα πρόγραμμα συνοχής δεν μπορεί να το λύσει αυτό το, ε, αυτό το ζήτημα. Ε, η κατάσταση επιδεινώνεται όλο και περισσότερο. Ε, θα σας πω ότι μόνο φέτος 200.000 εργαζόμενοι στην Ελλάδα δεν ανανεώσανε την άδεια για τα αυτοκίνητά τους γιατί δεν έχουν να πληρώσουν ε, το, το τέλος κυκλοφορίας. Είναι ψηλές οι τιμές στο πετρέλαιο με αποτέλεσμα η, η να έχει ξαναγυρίσει στην Αθήνα και αν η συνάντηση που ε, ε, προετοιμάζει η Ελληνική Προεδρία γινόταν το Φλεβάρι θα το νιώθατε άμεσα πόσο δύσκολες είναι αυτές οι συνθήκες και γενικότερα επειδή έγινε λόγος και για προγράμματα ανεργία των νέων και στήριξή του. Θέλω να ξέρετε ότι ορισμένα από αυτά που ήδη εφαρμόζονται στην Ελλάδα είναι με πολύ χαμηλού μισθού, ε, πεντάμινε συμβάσει, οι οποίε δεν ανανεώνονται και ε, μετά από αυτό οι εργαζόμενοι οι νέοι δεν έχουν το δικαίωμα να ε, γραφτούν στα γραφεία ανέβρεση εργασία, στα γραφεία ανεργία. Άρα δηλαδή αυτό το πρόβλημα θα υπάρχει και αν υπάρξει κάποια ε, ε, ανεμική ανάπτυξη, αυτή θα γίνει πάνω σε αντιλαϊκές και σε αντεργατικές ε, ρυθμίσεις. Αυτά που λέω δεν είναι θεωρία. Ξέρετε όλοι σας πάρα πολύ καλά ότι τα προγράμματα της, του Ταμείου Συνοχής μπαίνουν στην αιρεσιμότητα. Εάν δεν τηρούνται τα γνωστά κριτήρια θα υπάρχουν περικοπές και στα προγράμματα αυτά, πολύ περισσότερο που ο προσανατολισμός τους δεν εξυπηρετεί ε, τις αυξανόμενες ε, ανάγκες που υπάρχουν. Είτε μιλάμε για στέγαση, είτε μιλάμε για μεταφορές. Παραδείγματος χάρη, γιατί να μην υπάρχει δωρεάν μεταφορά των ανέργων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, γιατί αυτά τα προγράμματα, να μην, αυτά τα ποσά να μην χρηματοδοτούνται από τα ταμεία συνοχή, εφόσον υπάρχει τόσο μεγάλη ευαισθησία όσον αφορά του ανέργου. Ή αν θέλετε ένα άλλο θέμα, παραδείγματο χάρη που δεν να το κάνετε. Γιατί δεν χρηματοδοτείτε συστήματα τηλεθέρμανση. Και έχουμε τώρα την Ελλάδα και άλλες χώρες, ο καθένας να προσπαθεί να, να, να ζεσταθεί όπως μπορεί με τεράστια ε, πώς το λένε, ε, απώλεια και τεράστιες τιμές στην ενέργεια, στο πετρέλαιο κτλ. Γι' αυτό το λόγο εμείς είμαστε ε, ε απεσιόδοξοι. Πιστεύουμε ότι μόνο με ριζικές αλλαγές, μόνο με ανατροπή του καθεστώτος των μονοπωλίων θα μπορεί να υπάρχει μια ανάπτυξη που να εξυπηρετεί τις, ε, κοινωνικές ανάγκες. Γι' αυτό και κιόλας αγωνιζόμαστε για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όσο είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αυτό που θα εξυπηρετείται θα είναι τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και δεν θα μπορούν οι εργαζόμενοι να έχουν μια ανάπτυξη που να ανταποκρίνεται σε αυτό που ζητάνε. Thank you very much. We have two more... Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε δύο αγορητές που έχουν ζητήσει ακόμη το λόγο. Πρώτο πρώτο Γιάν Ολμπρίτ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε γιατί ξέρετε όλοι οι υπουργοί, όλες οι κυβερνήσεις ε, θα πρέπει να αναγνωρίζουν τι θα πει η Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε θα πρέπει κάπως να υπάρχει διαβούλευση επικοινωνία. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έκανε τη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι όλο ένα και περισσότερο ενδιαφέρεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή, την εκτέλεση. Ας πούμε, ολοκληρώσαμε αυτό το νομοθετικό πακέτο τη δέσμη μέτρων, αλλά εμεί θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας πριν το, το, το τέρμα, ούτως ώστε να έχουμε την ενημέρωση και το νέο κοινοβούλιο με σίγουρος θα είναι πάρα πάρα πολύ δυναμικό όταν έρθει η ώρα της ε, αναθεώρησης μετά τα 3,5 χρόνια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και γι' αυτό και είναι τόσο δύσκολη αυτή η προβληματική για την πολιτική της συνοχής. Τα είπαμε σήμερα, έχουμε τον έλεγχο. Δηλαδή, όλο ένα και μεγαλύτερο καθίσταται το ενδιαφέρον λόγω τη σημασία του. Και επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο εσεί δηλώσατε ότι ακόμα και σε σύντομη περίοδο θα υπάρξει αυτή η επαφή με την ελληνική προεδρία για την ε, όλη διαδικασία. Καταλαβαίνω, σήμερα ε, εκπροσωπείτε σε 28 χώρε και όχι την Ελλάδα, γιατί ακριβώς το, το, το, τα θέματα τα ιστορικά της Ελλάδος είναι ενδιαφέροντα, αλλά τώρα συζητούμε και ομιλείτε εσείς για όλη την Ευρώπη. Έχω μία ερώτηση όμως. Εσείς ως Προεδρία, τι, τι έχετε να πείτε όσον αφορά αυτά τα δεδομένα τα οποία σήμερα παρουσιάστηκαν από τον Γενικό Διευθυντή Ντέφα στην ε, συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ξεκίνησε να μιλάει για την πολιτική συνοχή λέγοντας ότι δεν έχουμε εκταμιεύσει και καταβάλει 16 δις τον Δεκέμβριο. Άρα το πρώτο εξάμεινο θα υπάρξει ένα τέτοιο πρόβλημα κενού στον προϋπολογισμό. Ποια είναι η θέση της ελληνικής προεδρίας, τι θα κάνετε στο Συμβούλιο με ε, αυτό το δεδομένο, σε έξι μήνες θα αλλάξετε τον προϋπολογισμό, θα κάνετε διορθωτική κίνηση. Εσείς τι θα κάνετε ως Προεδρία. Κύριε Φεραγκούτ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, και επίσης σας ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας εξηγήσατε και τις προτεραιότητες όλες που επισημάνατε όσον αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης, ε, το κείμενο αυτό το οποίο εμείς εγκρίναμε εδώ στην Επιτροπή μας και είπαμε ότι θα ολοκληρωθεί ο κανονισμό τον Μάρτιο χωρί καμία αμφιβολία. Πρόκειται κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η έκφραση τη ελεγγύη τη κοινοτική. Ε, Όντω θα υπάρξουν περικοπέ από τον προπολογισμό, αλλά εμεί αυτό το οποίο εδώ εγκρίναμε είναι κάτι το πιο ρεαλιστικό, κάτι πιο ρεαλιστικό από αυτά που γίνονται το 2005 και από πλευρά τη Επιτροπή και από πλευρά Γενοβούλου Γιατί έτσι ε, μπορούμε να πλαισιώσουμε, να, να κάνουμε κάτι για τι θεομηνίε, τι καταστροφέ, τι περιφερειακέ. Ε, εκεί δεν πρόκειται για κάτι το αόριστο του φλού, πρόκειται για ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και ποσοστό. Οπότε ε, τον ε, Δεκέμβριο τα ξαναείπαμε και τώρα θα έχουμε και συναντήσεις, αυτές που ονομάζουμε τριλόγους, οπότε θα πρέπει να σας διαβάσω το ότι χρειάζεται κάτι να γίνει, να εγκριθεί αυτό πριν το κοινοβούλιο διαλυθεί, μέχρι το Μάρτιο δηλαδή, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε την απαραίτητη ευελιξία, να μπορέσουμε στους τριλόγους να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία. Οπότε θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί, γιατί αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε αυτού του κανονισμού είναι να κάνουμε διορθωτικέ κινήσει και στη συνέχεια δεν να μπορέσουμε να κάνουμε την, την εφαρμογή, να χρησιμοποιήσουμε αυτό το, το, ταμείο και να έχουμε αυτό το 1% του ΑΕΠ και να πάει αυτό σαν αρρωγή στις ε, περιφερειακές ε, ε, θεομηνίες, φυσικές καταστροφές που λέμε και έτσι να καλύψουμε τις διάφορες περιφέρειες και επίσης να παρεκτείνω, παρατείνουμε τις, προθεσμίες ε, για την εκτέλεση, να υπάρξει δυνατότητα να γίνονται προκαταβολές ε, άπαξ και τέλος πάντων έχουν ξεκαθαριστεί όλα τα νομικά ζητήματα. Φαντάζομαι ότι τα τρία θεσμικά όργανα στο ίδιο μήκος κύματος και επίσης όσο γίνεται νωρίτερα να, να, να προσπαθήσουμε να κλείσουμε αυτό το θέμα και να έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια ε, σύντομα. Έχετε κύριε Υπουργέ τώρα το λόγο εσείς. Θα προσπαθήσω να είμαι συντομότατος. Πρέπει να τελειώνω σε 10 λεπτά. Γιατί πρέπει και εσείς να φάτε. Έχετε και άλλα πράγματα να κάνετε σοβαρότερα από το να ακούτε εμένα. Θα μιλήσω αγγλικά, δεν χρειάζεστε εσείς μετάφραση. Ε. Λοιπόν, καταρχάς, για αυτά που είπε ο Λάμπερτ Βανίστελ Ρόι και η Κωνσταντσα και άλλοι συνάδελφοι. για τις κατεξουσιοδότησης πράξης. Πρέπει να σας πω ότι ως Προεδρία έχουμε δώσει ένα μήνυμα ως προς τον κώδικα δεοντολογίας που προτείνουμε στα κράτη-μέλη και πρέπει αυτός ο κώδικς να εγκριθεί ως το δυνατόν συντομότερα. Βεβαίως υπάρχουν ακόμη προβλήματα άλυτα, αλλά νομίζω ότι με τη συνεργασία με την Κομισιόν, σε συνεργασία με την Κομισιόν θα ξεπεράσουμε αυτό τα εμπόδια γιατί αυτό θα ωφελούσε όλα τα κράτη-μέλη και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλύτερα βέβαια να μην υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, αλλά δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας mm. στα γεγονότα εξορισμού πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά και κατανοώ ότι οι χώρες μέλη το έλαβαν αυτό το μήνυμα γιατί είναι σημαντικό και για αυτά τα κράτη-μέλη. Χρειάζονται τα χρήματα από τα διαρθρωτικά ταμεία και γι' αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι τελικά θα επικρατήσει η κοινή λογική αυτό. είναι το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω τώρα ως Προεδρία. Όπως ξέρετε έχω και εγώ περιορισμούς. Και ζηλεύω λίγο γιατί εσείς έχετε την ελευθερία να εκφράζετε τις απόψεις σας χωρίς τα όρια που έχω εγώ ως εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Τώρα για, την εφαρμογή του κανονισμού, ο κύριος Γκοντμάνης αναφέρθηκε σε αυτό. Υπάρχουν βέβαια καθυστερήσεις. Μερικές χώρες μέλη υπέβαλαν τις προτάσεις τους, άλλες όχι. Είμαστε σε συνεχή επαφή με την Κομισιόν και πιστεύουμε ότι θα λυθεί και αυτό, Θα αντιμετωπιστεί. Βέβαια, για να υπάρξει έγκριση πρέπει πρώτα να έχουμε την πρόταση. Δεν είναι πρώτη φορά που υπάρχει αυτό το πρόβλημα των καθυστερήσεων δηλαδή. Θυμάμαι ότι το είχαμε και σε παραγωγούμενες προγραμματικές περιόδους, αλλά νομίζω ότι η Κομισιόν είναι αποτελεσματική και ο Επίτροπος Χάν θα έρθει νομίζω το απόγευμα εδώ, άρα μπορείτε να του το θέσετε. Και όπως είπα βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία για να το λύσουμε. Είναι πραγματικό πρόβλημα κύριε Γκουτμάνη μου. Τώρα στρέφομαι στα ελληνικά θέματα τον ρυθμό απορρόφησης κλπ. Είναι σαφές ότι αρχίσαμε πολύ άσκημα αλλά 18 μήνες μετά μετά τις εκλογές του 12 η Ελλάδα ως προς το ρυθμό απορρόφησης ήταν σε πολύ άσκημη θέση 18η ή 20η μεταξύ των 27 χωρών μελών παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα και στον τραπεζικό μας τομέα ρευστότητας, εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών. Κάναμε τρομακτική προσπάθεια και είπατε κι εσείς ότι τώρα είμαστε με τέταρτη ή πέμπτη, στην τέταρτη ή πέμπτη θέση. Για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο τώρα, τα πράγματα ήταν ακόμη χειρότερα πριν από μερικούς μήνες. Αλλά καλύψαμε το χάσμα και το κενό. Προς το Δεκέμβριο ο ρυθμός απορρόφησης για την Ελλάδα, για την συνολική δέσμη, έφτανε το 74% για το κοινωνικό δε ταμείο 62%. Δεν είναι και άσχημο. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και καλύτερος ρυθμός, αλλά... Αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη σας από πού αρχίσαμε. Τα διαρθρωτικά προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε, το πρόβλημα ρευστότητας, καθώς και την πρόοδο που επιτέχθηκε, που ήταν όχι να το περηφανευτώ, αλλά παραπάνω από σημαντική. Βέβαια ο αγώνας αυτός συνεχίζεται. Όχι μόνο για να έχουμε μια καλή εικόνα εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά γιατί αυτό είναι το πατριωτικό μας καθήκον. Τώρα, προς τον κύριο Βλάσακ θα ήθελα να πω για το κόσμο και το ορίζον. δεν είναι καθαρά δική μου δικαιοδοσία αλλά το Υπουργείο Παιδείας που καθώς και τεχνολογίας και έρευνας στην Ελλάδα που ασχολείται που είναι αρμόδιο. Ξέρω όμως ότι η Προεδρία ήδη έχει οργανώσει μία διάσκεψη για τα δύο αυτά προγράμματα στην Αθήνα και σχεδιάζουμε και άλλες εκδηλώσεις γιατί ένας από τους στόχους μας είναι να δράσουμε ως καταλήτης για να επιταχυνθούν οι εξελίξεις, να μην συνεχίσουν οι καθυστερήσεις σε αυτά τα δύο καινοτόμα προγράμματα. Για τον κύριο Αγκουράκη, γιατί θα ήταν λίγο άκομψο μεταξύ εκείνων να μιλάμε ε, ξένες ε, άλλες γλώσσες. Ή ε, όχι κύριε Αγκουράκη. Ε, εγώ σέβομαι τη θέση του κυρίου Αγκουράκη απολύτως. Αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας. Υπάρχουν διαφορετικές θέσεις μεταξύ των κομμάτων. Υπάρχουν οι εκλογές. Στη δημοκρατία ο λαός ακούει τις διαφορετικές απόψεις και αποφασίζει. Ε, σίγουρα έχουμε να κάνουμε μια πολύ δύσκολη δουλειά στην Ελλάδα. Έχουμε να χειριστούμε μια άνευ προηγουμένου κρίση. Ε, αυτή την ώρα έχουμε μια πρόοδο στο επίπεδο της δημοσιονομικής προσαρμογής. Ε, έχουμε το πέμπτο χαμηλότερο έλλειμμα σε όλη την ε, Ευρωζώνη. Έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, primary surplus, ξεπερνώντας τις προσδοκίες. Ε, στο επίπεδο των διαρθρωτικών αλλαγών ο OECD, ο ΩΣΑ μας κατατάσσει πρώτου στο Going for Growth Report σε όλα τα κράτη-μέλη του ΩΣΑ. Βεβαίως έχουμε μπροστά μας μια τρομερή άνευ προηγουμένου ενεργεία και μια πολύ μεγάλη εκτάσεως κρίση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ούτε θέλει να κρύψει κανείς κάτι, όμως νομίζω δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και φέτος περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί λένε ότι μετά από έξι χρόνια η Ελλάδα ε, θα περάσει από την ύφεση σε ρυθμούς ανάπτυξης. Και είναι στο χέρι μας όλοι μαζί να δουλέψουμε με σοβαρότητα και με εθνική ενότητα για να ξεπεράσουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι πρόβλημα που αφορά όλους τους Έλληνες. Ε, back to other questions. Λοιπόν, για να επανελθώ στα υπόλοιπα ερωτήματα. Ο κύριος Όλμπριχ αναφέρθηκε σε καθυστερήσεις πληρωμών, γεγονός, δυστυχώς. Νομίζω πως σχετίζεται με κάποια προβλήματα ρευστότητας ε, στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα προβλήματα που αφορούν τις σχέσεις ε, Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιόν τους τελευταίους μήνες. Είμαστε θύμα, εμείς ως χώρα εννοώ, των καθυστερήσεων αυτών και προσπαθούμε να μην ε, υπάρχει κάποιος αντίκτυπος στον προϋπολογισμό μας ε, λόγω των τεχνικών αυτών ζητημάτων και νομίζω πως ε, είμαστε κοντά στο να βρούμε μια λύση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην έχουμε αυτές τις συνέπειες αλλά το πρόβλημα αυτό δεν έχει σχέση με την Προεδρία έχει σχέση με το παρελθόν το κληρονομήσαμε και νομίζω πως ε, σύντομα θα το αντιμετωπίσουν οι υπηρεσίες της ε, Κομισιόν. Και τέλος. Κύριε Στέρας, ως ε, Προεδρία οργανώσαμε ήδη δύο συναντήσεις τον Ιανουάριο το επίπεδο του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Λεγγύης και προγραμματίζουμε μια τρίτη συνάντηση 31 Ιανουαρίου στο τέλος του μήνα και προσπαθούμε να βρούμε κάποιον κοινό παρονομαστή με τα άλλα κράτη-μέλη. Βεβαίω, αντιλαμβάνεστε, είναι προφανές πως έχουμε κάθε λόγο να προωθήσουμε την υιοθέτηση του νέου κανονισμού και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμά μας πρέπει να σας πω πως ο στόχος μας η φιλοδοξία μας είναι να ξεκινήσουμε τριλόγους ή δυνατόν τα μέσα Φεβρουαρίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμά μας και ελπίζω σε συνεργασία με τα άλλα κράτη-μέλη και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιμείνουμε σε αυτό. Αυτά είναι τα σχόλιά μου. 12 λεπτά ήταν η παρέμβασή μου. Χάρηκα που σας ξαναείδα. Είμαι στη διάθεσή σας και θα συνεχίσουμε βεβαίως ε, την επαφή. Ε, θα πρέπει να είναι ελληνική η Προεδρία γιατί πρέπει να κάνετε τη δουλειά εξαμήνου σε τρεις μήνες. Ναι, πράγματι, θα γίνουν όλα στην αρχή, λέει ο κ. Φατζητάκης, αλλά είπα, είμαστε καταδικασμένοι να επιτύχουμε. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ό,τι χρειάζεστε, λοιπόν, θα σας στηρίξουμε ειδικά για την πολιτική συνοχή. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία.